domnul președinte ședința este reluată. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Ε, τα συνοπτικά πρακτικά έχουν ε, διανεμηθεί, ε, διατίθεται, καθώς επίσης και τα κείμενα που εγκρίθηκαν χτες, τα χτεσινά συνοπτικά πρακτικά, και αν δεν έχετε σχόλια θεωρούνται εγκεκριμένα. Ωραία. Προχωρούμε λοιπόν στο πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης για το απόγευμα, που είναι η έκθεση κυρίας Ρης, με θέμα τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Κυρία Ρης, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ακόμα έφτιαχνα τι σημειώσει μου. Ε, κύριε Αντιπρόεδρε Τίμερμαν, σα βλέπω εκεί. Είσαι και εσά, κύριε Επιτρόπε, κύριε Βέλα. Ε, θα ήθελα λίγο να κάνω μια ιστορική αναδρομή εδώ. Θυμάστε εκείνη τη βραδιά 18 προς 19 Δεκεμβρίου τη νύχτα στο τριμερή διάλογο 20 ε, χρόνια είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αν έχω ζήσει τριμερείς διαλόγους ε, και αυτός ο τριμερής διάλογος είπε όχι στα πλαστικά μιας ε, χρήσεως 12,5 ώρες μαραθώνιες διαπραγματεύσεις χρειάστηκαν με το Συμβούλιο για να γεννηθεί η πιο φιλόδοξη νομοθεσία και να είμαστε υποδειγματικοί δεν είχαμε άλλη επιλογή παρά να ηγηθούμε στη μάχη αυτή Δεκάδες φορές χρειάστηκε να παρέμβω σε ακροάσεις στην Επιτροπή, στην ομάδα, στην Ολομέλεια. Θύμισα τα αριθμητικά στοιχεία, τις εικόνες, την τραγική κατάσταση των ωκεανών μας, αλλά και στην Ευρώπη. Τα πλαστικά δηλητηριάζει τις θάλασσές μας, ε, σκοτώνει ε, τα όντα που ζουν στη θάλασσα και τελικά απειλεί εμάς που είμαστε στο τέλος αλυσίδας. 70% του συνόλου των ε, σκουπιδιών στη θάλασσα είναι πλαστικά μιας χρήσης και μαζί με τα αλλιευτικά εργαλεία. Νύψαμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία με την Αυστριακή Προεδρία και είναι πολλές συνήκες που αξίζει να υπογραμμίσουμε. Πρώτον, ε, η επέκταση του καταλόγου των πλαστικών μιας χρήσης που ε, θα απαγορευτούν μετά από δύο χρόνια. Το 2021 είναι αύριο. Ε, τα πλαστικά πιάτα, ε, ε, μαχαιροπύρουνα, αναδευτήρες, μπατονέτες και τα, οι, συσκευ... οι πλαστικές συσκευασίες, όξο και φρίγκολίτ. Δεν ήταν καθόλου εύκολο αυτό απέναντι σε ένα διστακτικό συμβούλιο. Ε, το καθεστώς ε, της ε, ευθύνη του παραγωγού. Ο πληρώνει, έχει διευρυνθεί και πλέον βρίσκεται στο κέντρο της νομοθεσίας μας. καταφέραμε η καπνοπαραγωγή να είναι υποχρεωμένη να χρηματοδοτούν τη συλλογή, την απορρίπανση και την ανακύκλωση των αποτσιγάρων και αυτό από τον Ιανουάριο 2023, ένα χρόνο νωρίτερα από τους υπολείπους